Νομίζω καλό θα ήταν να αρχίσουμε σιγά σιγά. Η άγκριση της ημερήσιας διάταξης. Διαφωνείτε. Τα πρακτικά εγκρίνονται και αυτά. Προχωρούμε. Μερικές ανακοινώσεις. Μεταδίδεται ε, στο διαδίκτυο απευθείας η συνεδρίαση. θα δείτε και ε, τα όσα έγιναν στις 18 Οκτωβρίου ένα σημείωμα στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά για τα όσα διαμήθησαν με τον κοινωνικό διάλογο. Ε, οι συντονιστές θα συνεδριάσουν αμέσως μετά τη συνεδρίασή μας. Το σημείο που σας αναφέρω λέγεται 18 κάθετος 2011. Uh, I think it's too close. Um, uh, θα Έλεγα λοιπόν ότι οι συντονιστές θα συνεδριάσουν αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίασης, ό,τι ώρα τελειώσει η συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας. Ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν στο πρώτο θέμα στη μέση διάταξη, η διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η συγγήτρια είναι η κυρία Εύελιν Ρέγνερ, αλλά θα την αντικαταστήσει η κυρία Στάινοκ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Ρέγνερ με παρακάλεσε να σας παρουσιάσω τη γνωμοδότησή της, γιατί σήμερα κολλείεται. Η κυρία Ρέγνερ θέλει να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τακτική της ε, ε, ε, κανονικά ε, υπάρχει μια διαδικασία ε, που ακολουθείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί μια διαφορετική με τη νέα διατύπωση που δεν αναποκρίνεται στις απαιτήσει. Στην αναδιατύπωση δηλαδή. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επεκταθεί η εφαρμογή, το πεδίο εφαρμογή και σε πολίτες τρίτων χωρών και διευρύνεται ε, πολύ. Ε, αυτό λοιπόν είναι αναδιατύπωση της οδηγίας ε, και όχι νέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να περιορίζει εκ των προτέρων το δικαίωμα των βουλευτών, ούτε να ορίζει τι πρέπει να αλλάξει και τι επιτρέπεται να αλλάξει. Γι' αυτό οι τροπολογίες της κυρίας Ρέγνερ θα πρέπει να γίνουν δεκτές, είναι απαραίτητες από νομικής απόψεως. Να σας πω γιατί γνωρίζουμε ότι η Ρώμη 2, ο κανονισμός αυτός, ορίζει ποιο το δίκτυο εφαρμόζεται. Ε, ο κανονισμός Βρυξέλλης 1 μας λέει μόνο σε ποιο ε, μέρος θα γίνει η ε, διαδικασία αυτή, ενώ θα πρέπει οι δύο κανονισμοί αυτοί να συνδυάζονται. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό Ρώμη 2, εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας όπου υπάρχει η διένεξη. Ας πούμε, αν γίνει απεργία στη Σουηδία, εφαρμόζεται το σουηδικό δίκτυο, δίκαιο συγγνώμη, στο διακανονισμό. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να ψηφίσουμε τις ε, τροπολογίες της κυρίας Ρέκνερ. Θα πρέπει ε, ε, ο διακανονισμός και πύλης των διαφορών να γίνεται στη χώρα όπου έγινε η απεργία. Θα ήταν ε, παράλογο ένα βουλγαρικό δικαστήριο να αποφαίνεται για μια απεργία που γίνεται στη Σουηδία εφαρμόζοντας μάλιστα το σουηδικό δίκαιο. Ιδιαίτερα το κοινωνικό δίκαιο και το εργατικό δίκαιο που είναι σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των κρατών μελών. Γι' αυτό ε, ε, το βουλγαρικό δικαστήριο θα εφήρμοζε αυτό το δίκαιο. Δεν μπορεί κανείς να με πείσει ότι όλα τα δικαστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει η κυρία Ρέγνερ, γνωρίζουν το εργατικό δίκαιο όλων των κρατών μελών. Γι' αυτό ζητεί, ε, τα όσα ζητεί η κυρία Ρέγνερ. Στο άρθρο 85 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι δεν ε, επηρεάζει ε, τις εργατικές διαφορές αυτή η πρότασή της. Κανονικά θα πρέπει να λέει ο κανονισμός ρητά πού θα γίνεται η διαδικασία. Κανονικά θα πρέπει να είναι στη χώρα που θα γίνει τη απεργία. χωρίς ε, να χρειάζεται κάποιος να κρίνει το δίκαιο της χώρας αυτής. Και τα οικία δικαστήρια γνωρίζουν καλύτερα το δίκαιο της χώρας, θα πρέπει να είναι παραδεκτές αυτές οι διακασίες και κατά τα άλλα κυρία Ρέγνερ παρακολουθεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει γιατί ε, δεν ε, αναγνωρίζει στους βουλευτές το δικαίωμα να υποβάλουν προτάσεις τροποποίησης. Ελπίζω να ανοίξει αυτό τα μάτια και σε άλλους συναδέλφους των πολιτικών ομάδων και να υπερψηφίσουν τις δικές μας τροπολογίες. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι για μας τους βουλευτές το δικαίωμα ε, νομοθετικής δραστηριότητας. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Άλλοι αμιλητές για αυτό το θέμα. Uh, well... Ε, όχι. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, κάποιος ζητάει το λόγο. Α, ο κύριος Μπαλτασάρη, συγγνώμη. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ κατανοώ απόλυτα τις δυσκολίες μεταξύ των οποίων κινήθηκε η συνάδελφος ε, ε, Ρέγνερ και προσπάθησε φυσικά να κάνει όσο γίνεται καλύτερη δουλειά. Όμως κατά τη γνώμη μας πολλές από τις ε, τροπολογίες της είναι στην ουσία νέα στοιχεία που είναι ασύμβατα με το σχέδιο αναδιατύπωσης σε κάποιες από τις ε, τροπολογίες ε, μπαίνει στην ουσία του συστήματος με την εισαγωγή νέων ε, κανόνων και διαδικασιών που ωστόσο δεν συνοδεύονται από την κατάλληλη, την επαρκή αξιολόγηση αντίκτυπου. Πρόκειται για μέτρα τα οποία θα τροποποιούσαν σε σημαντικό βαθμό το σύστημα που ισχύει μέχρι σήμερα αλλά που κατά κανένα τρόπο δεν έχουν αξιολογηθεί Και πιστεύω λοιπόν ότι αν και καταλαβαίνω ότι οι προθέσεις της εισηγήτριας ήταν ε, θεμητές και κατανοητές, αυτές οι απόπειρες βελτίωσης ε, κατά τη γνώμη μας δεν είναι οι κατάλληλες. Άρα λοιπόν, Τόσο όσον αφορά την συμβατότητα των προτάσεων αλλά και των τροποποιήσεων που, που υποβάλλονται, εμείς δεν βρίσκουμε σημείο σύγκλησης. Η δικιά μας εκτίμηση είναι λοιπόν αρνητική και άρα η ψήφος του ΕΛΚ δυστυχώς δεν θα είναι υπέρ αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ άλλος. And Mrs. Yes. Uh, Cecilia Wikström could be not be here today. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Σεσίλια Βίξτρομ απουσιάζει γιατί κολλείται και επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω μερικά σχόλια από πλευράς της για αυτό το σημαντικό θέμα. Καλωσορίζει η Σεσίλια την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής και αποφάσεις ε, να ε, την ακολουθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Σήμερα όμως υποστηρίζουμε μόνο μερικές τροπολογίες. Μεταξύ αυτών ε, η τροπολογία της εισηγήτριας να προσθεθούν και οι απεργίες στη δικαιοδοσία για να μην υπάρχει ε, ένα shopping, μια ε, διακριτική επιλογή, όπως λέει η τροπολογία 2. Επίσης, το δικαστήριο που θα αποφαίνεται θα πρέπει να είναι δικαστήριο κράτους ε, που γίνεται η απεργία, ε, όπως ορίζει η τροπολογία 14. Σε ό,τι αφορά όμω το ε, άρθρο 19.2, όπου μπορεί να γίνει, κατατεθεί αγωγή κατά ενός εργοδότη, εμείς καταψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ. Η κυρία Στάιρουκ θέλει να προσθέσει τίποτα. Όχι. Αν δεν έχουμε τίποτα άλλο, η ψηφοφορία θα γίνει αργότερα εντός της σήμερα όπως γνωρίζετε και προχωρούμε μέσω στο επόμενο θέμα. Ε, υποθέτω ότι θα παρευρίσκεται βέβαια ο εισηγητής ή η εισηγήτρια. Είναι η έκθεση της Σιλβάνα Ράπτη, αναθεώρηση ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Η κυρία Ράπτη. Την αντικαθιστά κανείς. Είναι καθοδόν. Ο κύριος Σέρκας. Κάποιο μικρό πρόβλημα μάλλον θα έχει η κυρία Ράπτη. Εδώ ήταν στη συνεδρίασή μας, είναι στο Κοινοβούλιο. Αν μπορούσαμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα και στο μεταξύ να την ψάξουμε, γιατί το πρώτο θέμα τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα και την ξεπεράσαμε εμείς ε, από ταχύτητα. I'd Αν έρθει σε λίγα λεπτά, θα προτιμούσα να περιμένουμε. Γιατί μετά δεν θα είναι εδώ η αρμόδια της επόμενης έκθεσης. Καλό θα ήταν περιμένουμε λίγο την κυρία Ράπτη. Κάποιος μου λέει ότι είναι καθοδόν και θα φτάσει σε ένα-δύο λεπτά. Στην περιμένουμε. Άλλες ανακοινώσεις δεν έχω να κάνω. Ε, τι να κάνω, δεν μπορώ να μιλάω και ώρες για το ίδιο θέμα. Θέλετε να σα πω τίποτα άλλο. Ε, μην φύγετε, απλώ <laughs> έτσι να πούμε τίποτα άλλο. Um, okay, we'll just have a one or two minute break. Ας περιμένουμε ένα-δύο λεπτά. Oh, η κυρία Ράπτη ήρθε. Ας της αφήσουμε λίγο χρόνο μέχρι να καθίσει και θα ξεκινήσουμε. Είναι η έκθεση λοιπόν της κυρίας Ράπτη για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Ε, μιλάμε για μια γνωμοδότηση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Όπως όλοι ξέρετε, η κύρια επιτροπή είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Σε μας πέφτει το βάρος να δώσουμε την δική μας ματιά, τη δική μας γνώμη για το πώς η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα μπορέσει να βοηθήσει στο επίπεδο της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων. Το πρώτο που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω τους συναδέλφους τους Σκιώδης. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και βοήθησαν στο να γίνει η γνωμοδότηση αυτή ε, πραγματικά ακόμα πιο σταθερή, ακόμα πιο ελπιδοφόρα είναι ιδιαίτερη συγκυρία στην οποία γίνεται αυτή η γνωμοδότηση και μιλάω βέβαια για την αραβική άνοιξη παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας περιλαμβάνει χώρες που βρίσκονται ε, και στα ανατολικά σύνορα της ευρωπαϊκής ένωσης αντιλαμβάνεστε ότι λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης που επικρατεί αυτό τον καιρό στην περιοχή της Βορείου Αφρικής δίνουμε ε, βαρύτητα στην, στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και στα επίγοντα ζητήματα των χωρών αυτών. Κατατέθηκαν συνολικά 66 τροπολογίες ανάμεσα σε αυτές είναι και δικές μου τροπολογίες γιατί όπως ξέρετε υπάρχει ο περιορισμός των λέξεων στην σύνταξη μιας γνωμοδότησης και κατά συνέπεια προσθέτουμε με τροπολογίες μετά. Οι περισσότερες τροπολογίες ακολουθούν τη φιλοσοφία της γνωμοδότησης, την κάνουν πληρέστερη και γι' αυτό τις υπερψηφίζουμε προσπάθησα να ενσωματώσω πολλέ από τις τροπολογίες όσο περισσότερες γινόταν στις συμβιβαστικές τροπολογίες. έχουμε καταλήξει σε εννέα συμβιβαστικές τροπολογίες. τα βασικά σημεία πάρα πολύ σύντομα για να μην σας κουράζω είναι τα εξής οι απαραίτητες δομικές οικονομικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην απασχόληση και στην κοινωνική προστασία δεύτερον η ενίσχυση διοικητικών ικανοτήτων και των κοινωνικών εταίρων με τη στήριξη από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τρίτον να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως η ανισότητα των φύλων η υποαπασχόληση των νέων και η παιδική εργασία. Τέταρτον, να υπάρχει έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης όπως και της κυκλικής κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφύγουμε την ενδεχόμενη διαρροή εγκεφάλων από τις χώρες αυτές. Πέμπτο και τελευταίο, οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με προϋποθέσεις βέβαια και η προϋπόθεση είναι να ακολουθούνται οι θέσεις μας ιδιαίτερα σε σχέση με τις πολιτικές απασχόλησης. Εδώ βάζω τελεία και ε, μάλλον πριν βάλω ε, τελεία υπάρχει μία τροπολογία. Η τροπολογία 37. Η τροπολογία 37 ε, μιλάει για τον ελάχιστο μισθό. Μία προφορική τροπολογία να προσθέσω εδώ και να βάλουμε το εξής το λέω στα αγγλικά reminds about the necessity to... Υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να εξασφαλιστεί ότι ο κατώτερος μισθός παρέχει επαρκές επίπεδο διαβίωσης για τους εργαζόμενους ε, the minimum wage according to national practices. Έτσι νομίζω ότι θα είμαστε α, δίκαιοι και θα βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο τις χώρες αυτές. Εδώ τώρα βάζω την οριστική τελεία. Και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you. Um, uh, Ms. Elizabeth Moranchati. Mrs. Moranchati. Merci, Madame. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. η συγκεκριά μας για το θέμα κατόρθωσε να συμπεριλάβει το θέμα απασχόλησης και κοινωνικών θεμάτων μαζί με μια εξωτερική προοπτική, προοπτική εξωτερικής πολιτικής όσον αφορά την πολιτική γειτονία. Και νομίζω για την επιτυχία της πολιτικής γειτονία είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη και το κοινωνικό οικοδόμημα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί και σε πολιτικό επίπεδο. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ράπτη, διότι έδειξε, μεγά έδειξε ανοιχτό πνεύμα ε, και άνοιγμα για επικοδομητικό διάλογο με όλες τις πολιτικές ομάδες, τουλάχιστον ομιλώ εκ μέρους του ΕΛΚ για να μην υπάρχουν πλέον ορισμένες παρανοήσεις που υπήρχαν αρχικά και ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις ε, που ε, μας οδηγούν όλους σε μια συνεκτική αντιμετώπιση της γνωμοδότησης όπως μας προτείνεται. Χαιρετίζω λοιπόν το θετικό πνεύμα και νομίζω ότι μόνο επικοδομητική δουλειά ακριβώς σαν αυτή που έχει γίνει εδώ μπορεί να μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε πραγματική συμφωνία και σε αποτελεσματική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την κυρία Ράπτη και το ΕΛΚ θα ψηφίσει υπέρ τη έκθεση αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Μου λένε να περιμένω. Όχι, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you. Ευχαριστώ πολύ jelko kacin kes on äh, alde variraportöör Ευχαριστώ. Ελίκο Κότσιν που είναι σχεδόν συζητητής ε, από του φιλελευθέρους. Ζητά συγγνώμη που δεν ε, είναι παρόν σήμερα. Και θα ήθελα να μεταφέρω το μήνυμά του. Ο θα ήθελε καταρχήν να ευχαριστήσει την κυρία Ράπτη για τη συνεργασία και χαίρομαι διότι και η κυρία Ράπτη θεωρεί ότι ήταν πολύ καλή η συνεργασία την οποία είχαν. Χαιρετίζουμε αυτή την γνωμοδότηση, ιδίως ε, με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει στη Βόρεια Αφρική. Και ο σκιώδης συζητητής μας είναι ικανοποιημένο διότι περιλαμβάνεται και η ανατολική διάσταση, διότι εκεί υπάρχουν διαφορετικές τάσεις. Οι προτάσεις μας δεν αλλάζουν τη γνωμοδότηση, απλώς την διευρύνουν. Εάν εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τις γειτονικές χώρες, ε, αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει στις πολιτικές που έχουν σχέση με το εργατικό δίκαιο σε αυτές τις χώρες και έχει σχέση και με τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης αυτό. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερος ε, διότι η Συγκήτρια συμφώνησε να ε, συμπεριληφθεί η μεσογειακή διάσταση ένα θέμα στο οποίο έλαβε θέση και το Κοινοβούλιο στη γραπτή δήλωση του Σεπτεμβρίου. Υποστηρίζουμε τη γνωμοδότηση αυτή και θα ψηφίσουμε υπέρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κανεί άλλο το λόγο. Κυρία Ράπτη, θέλετε εσεί να λάβετε το λόγο. Ε, ξέρετε, ένα πολιτικό όταν του δίνουν το λόγο πάντα λέει ναι. Ε, έτσι και εγώ παίρνω για μία ακόμη φορά το λόγο. Ε, ευχαριστώ τους συναδέλφους και εύχομαι πάντοτε να έχουμε τέτοιου είδους συνεργασίες για να μπορούμε να βοηθούμε και, τον, και τους ευρωπαϊκούς λαούς αλλά και τους γειτονές μας. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ και η ψηφοφορία όπως γνωρίζετε θα γίνει σήμερα αργότερα. Πηγαίνουμε πολύ νωρί, δεν ξέρω αν μπορέσουμε να κάνουμε τελικά τι ψηφοφορίε νωρίτερα. Θα πρέπει να συμφωνήσουν οι πολιτικέ ομάδε για το αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε το πάντως, γιατί πρέπει να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει ψηφοφορία λίγο νωρίτερα. Και περνάμε στην έκθεση Καρή Μαντέλη για την ενδιάμεση αναθεώρηση τη Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2007 με 2012 σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Κυρία Ντελή. Merci, ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τρίτη φορά συζητάμε για αυτή την έκθεση. Έχουμε ήδη παρουσιάσει τις διάφορες τροπολογίες, πάνω από 200 ήταν. Ανάμεσα στους ε, σκιώδες εισηγητές είχαμε μια πρώτη συνεδρίαση που κατέληξε σε κάμια εικοσαριά συμβιβαστικές και μάλιστα θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά για την ποιότητα των, της συνεργασίας με τους κοιόδης εισηγητές είχαμε έναν διάλογο επί της ουσίας. Έναν, μια πραγματική συζήτηση που επέτρεψε να αρθούν οι αμφισημίες και να προχωρήσουμε πολύ πιο πέρα από αυτό που είχα αρχικά την πρόθεση. Πολύ ειλικρινά λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των σκιωδών εισηγητών για την αποτελεσματικότητά τους και για την ικανότητα καθώς και το κέριο χαρακτήρα των τροπολογιών τους. Σήμερα έλαβα την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΝΒΗ για την έκθεσή μου. Δεν την έχω ακόμα μελετήσει. Και φυσικά και θα το πράξω με μεγάλη προσοχή. Άρα λοιπόν σήμερα εξακολουθούμε να είμαστε στο θέμα των συμβιβαστικών τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ο κ. Πάρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ ευχαριστώ για την εργασία της εισηγήτρης και για την εκδοχή των συμβιβαστικών τροπολογιών που τη λάβαμε την Παρασκευή είναι εκδοχή, λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές και τις διεκδικήσεις που είχαμε αναφέρει κατά τη διάρκεια της συνάντησης των σκιωδών εισηγητών. Μια συνάντηση όπου στηρίζω και την ε, γνώμη της, ε, της κυρίας Νταλή και κυρίως για αυτές τις ε, νέες συμβιβαστικές, κυρίως αυτήν για το στρες στην εργασία, την ε, καθώς και την ν για τις μη δηλωμένες δραστηριότητες. Επίσης, το, όσον αφορά την συμβαστική β, με την έκδοχη η συγγήτρια μπόρεσε να βρει να, να, μια πρόταση πιο ισορροπημένη και ωστόσο κάποιες εξηγήσει για την συμβιβαστική WW όπου είχαμε διάφορες εξηγήσει και ίσως η συγκήτρια εκεί θα μπορούσε να αναλύσει κάπως περισσότερο αυτήν τη συμβαστική W για να έχουμε όλη την ίδια ερμηνεία. Ε, ε, Ευχαριστώ κυρία Ράπτη. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Καρή Μαντελή, η οποία αποδεικνύεται μια πάρα πολύ καλή μαγείρισα εντός εισαγωγικών. Μαγείρεψε εντός εισαγωγικών πάρα πολύ καλές συμβιβαστικέ συμβιβαστικές τροπολογίες και την ευχαριστώ γι' αυτό. Και αν μπορώ να κάνω άλλο ένα λογοπαίγνιο, οι τροπολογίες που μας παρουσίασε είναι και υγιείς και ασφαλείς ε, θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και θα ήθελα απλώς να τονίσω μερικά πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται συνεχώς και όσο περισσότερο ακούγονται τόσο καλύτερο κάνουν. Ε, πιστεύω ας πούμε ότι οι σωστές συνθήκες εργασίας πρέπει να είναι κριτήριο για την ανάθεση έργων ώστε να ανταμείβονται οι εταιρείες που λειτουργούν με πραγματικά συνθήκες κοινωνικής ευθύνης. Ε, το δεύτερο είναι ότι πρέπει να προσπαθούμε να προλαμβάνουμε μέσα από την καινοτομία ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια. Ε, είναι επίσης πολύ σημαντικό να εντοπίζουμε νέους κινδύνους στην εργασία οι οποίοι προέρχονται από νέα υλικά. Να αξιολογούμε επαγγέλματα ε, βεβαίως υπερθεματίζουμε την πρόταση της Καρίμας για μια οδηγία που αφορά το στρες. Ε, ενισχύουμε το αίτημα για ειδική μέρημνα, να γίνονται καλές χρήσεις, να γίνεται καλύτερη χρήση των στατιστικών στοιχείων, να έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους για την αξιολόγηση των κινδύνων, να προστατεύονται όλοι εκείνοι οι εργαζόμενοι που καταγγέλουν παράνομες ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Ε, και τέλος θα πρέπει οι τιμές και οι δείκτες που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία να μην μειώνονται να μην πηγαίνουν προς τα κάτω κάθε φορά που προσπαθούμε να απλοποιήσουμε την νομοθεσία μας. Εδώ βάζω μία τελεία και λέω άλλο ένα ακόμη ευχαριστώ στην Καρίμα. Thank um, Σας ευχαριστώ, κυρία Οβίρ. Θέλετε να μιλήσετε εξ ονόματος του σκιώδης Στην πρώτη μου ομιλία τα είπα ήδη αυτά που έπρεπε να πω εξ ονόματος της, ε, του σκιώδους εισηγητού, οπότε δεν θέλω άλλο το λόγο. Ο κύριος Μάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν κοιτάξουμε αυτές τις συμβιβαστικές προτάσεις που ψηφίστηκαν, που συμφωνήθηκαν, φαίνεται ότι άξιζε το κόπο να συνεννοηθούν όλοι και όλοι οι συγητές για να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός Β, για παράδειγμα, που έχω βάλει και εγώ το χεράκι μου εκεί για τις ρυθμίσεις της ε, κυριακάτικης εργασίας. Να μην γίνει κανονική εργάσιμη μέρα και η Κυριακή ε, με τεράστιες ε, δράσεις πολίσεων κτλ. Νομίζω καλά κινηθήκαμε εκεί και επιπλέον άτυπες μορφές εργασίας, η μερική απασχόληση αυξάνονται με ταχύτητα τους ρυθμούς και αυτό δεν θα πρέπει απλώς να τα περνάμε στον τούκου, να έχουμε σαφείς ε, δομές και να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι. Σε αυτή λοιπόν τη συμβιβαστική τροπολογία δε καλά κάνουμε και λέμε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τι αναφέρεται εκεί Πρέπει να επικρατήσει για ασφάλεια να το διευκρινίσουμε. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε και μπορούμε σε πνεύμα συνεργασίας να προχωρήσουμε. Ότι γίνονται αλλαγέ φαίνεται σε διάφορα κράτη αυτό. Έχεις τους χρόνους εργασίας, ας πούμε, ή πώς Ε, μεταφράζει το κατώτατος μισθός ή το κατώτατο όριο. Όλα αυτά τα όρια είναι πάρα πολύ ασαφή και ρευστά. Να δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα ή το επόμενο Σαββατοκυριακό. Να το καταλάβουν και οι εργαζόμενοι ότι γίνεται πρόοδος. Ε, φύγαμε από τα ε, μαξιμαλιστικά που θέλαμε τις μέγιστες απαιτήσει. γεννηθήκαμε λίγο, αλλά θα πρέπει τελικά να ε, πληρώνονται δίκαια όσοι εργάζονται, να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τι γίνεται και νομίζω τελικά θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση της Επιτροπής μας. Um, uh, Ευχαριστώ. Να ζητήσω συγγνώμη που δεν είναι εδώ. Ο κύριος Κρόιτς. Ε, Κρότσμαν. Ε, έχουμε κάποια προβλήματα ακόμα με κάποιες από τις τροπολογίες, ιδιαίτερα όσον αφορά κάποια νομοθετικά ζητήματα, όπως γνωρίζετε. Η συμβιβαστική W αναφέρθηκε από τον κύριο Μπάρκ και έχουμε ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή με αυτή τη συμβιβαστική. Επειδή δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι τι σημαίνει, αλλά φαίνεται να στρέφεται προς ένα νομοθετικό μέσο. Αν αυτό διευκρινιστεί θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε. Αλλά πέρα από αυτό, Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να το δουλέψουμε κάπως περισσότερο και να κάνουμε και κάποιες προσαρμογές σε αυτές τις τροπολογίες. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν που ο κύριος Κρόιτσμαν δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Να δώσω και πάλι το λόγο στην Καρίμα Ντέλη για να συνοψίσει. Σα Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ είμαι αρκετά ικανοποιημένη γιατί όλοι είστε στο ίδιο μήκο κύματο με μένα. Έτσι θα έχουμε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο κείμενο και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Ε, σημείωσα τα αιτήματά σας και ιδιαίτερα αυτή τη περίφημη συμβαστική W, που δημιουργεί απορίες. Εγώ θα είμαι σαφής. Η συμβαστική W θέλει να κάνει ένα κατάλογο επαγγελματικών ε, ασθενειών. Αυτός ο κατάλογος θα είναι υποχρεωτικό. δεσμευτικό. Είναι ένα αίτημα που προκύπτει από τους κοινωνικού εταίρου. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η γνωμοδότηση με, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος θα με οδηγήσει στο να ξαναγράψω αυτή την συμβαστική. Όμως θέλω να με σαφής για αυτήν. Εδώ ζητάμε έναν κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών που πρέπει να είναι δεσμευτικός. και τα λοιπά, να ευχαριστήσω τους, ε, άλλη μια φορά τους σκιώδεις εισηγητές και να συνεχίσουμε έτσι ωραία και για το υπόλοιπη συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντέλη. Ντελή. Και με, να σας πω πότε θα ψηφίσουμε προβλέπετε στις 23 Νοεμβρίου η υιοθέτηση στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης και να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι for Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συντερισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων. Η συγητής είναι ο κύριος Γκεγκούλτ των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν για τις τροπολογίες που είχατε την καλοσύνη να υποβάλλατε, 68 τροπολογίες έχουμε και οι περισσότερες επιβεβαιώνουν τη γενική γραμμή που προσπαθούσα να προτείνω κι εγώ στην έκθεσή μου. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία αποτελεί μια θετική εξέλιξη αλλά χρειάζεται να ε, τηρούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων ε, και τα δικαιώματα των υπαλλήλων στο ε, συνεταιρίζεστε και τονίζουμε επιπλέον και την ανάγκη βελτίωσης αυτής της νομικής μορφής και παράλληλα χρειάζονται και συμπληρωματικά μέτρα που πολλές φορές έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υποστηρίξουμε τον συνεταιριστικό τομέα και τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας γενικότερα. Τις περισσότερες τροπολογίες μπορώ να τις δεχτώ και αρκετές τροπολογίες αφορούσαν το ίδιο σημείο. Ήταν παρόμοιες δηλαδή τροπολογίες, οπότε διαμορφώσαμε συμβιβαστικές τροπολογίες και θα γίνει μια συνάντηση των σκιωδών εισηγητών επ' αυτού. Δεν θέλω τώρα ε, να, να σας ε, σπαταλήσω το χρόνο. Καλύτερα να ακούσω τι έχετε να πείτε. Έχουμε λάβει επίσης και γνωμοδότηση από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και από την Επιτροπή Γυναικών. Είναι η δεύτερη Επιτροπή. Η Επιτροπή Γυναικών όμως έχει ένα σχέδιο γνωμοδότησης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ψηφοφορία. Ακόμη περιμένουμε λοιπόν τη γνωμοδότηση της δεύτερης Επιτροπής. Περιμένω πάντως τα σχόλιά σας και στη συνέχεια στη διάθεσή σας να απαντήσω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους υποβάλλατε τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ, Μάριαν Χάρκινγκ, για το ρόλο των εργαζομένων στους ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που καθυστέρησα και για την προηγούμενη έκθεση είχα κάτι, αλλά θα το δώσω στην Καγιμαντελή γραπτός. Όσον αφορά την έκθεση αυτή τώρα, η Νάντια Χίρς ε, είναι σκιώδη συγγήτρια ε, εκ μέρου ε, των φιλελευθέρων και δεν μπορούσε να είναι σήμερα παρούσα και μου ζήτησε να κάνω τα εξή σχόλια. Καταρχήν, ευχαριστεί τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Ευχαριστεί και τον εισηγητή για τις προσπάθειες που έκανε μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές για να βρουν μια κοινή γραμμή. Λέει ότι η ανάγκη μια έκθεση σχετικά με τις συνεταιριστικές εταιρείε είναι περισσότερο επίγουσα από ποτέ γιατί οι συνεταιριστικές εταιρείε μπορούν να καλύψουν το κενό μεταξύ του δημόσιου τομέα και της ιδιωτικής οικονομίας. Συμφωνεί με τις περισσότερες τροπολογίες του εισηγητού που τονίζουν τα σημεία της έκθεση σχετικά με το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη με την τροπολογία 23. Θεωρεί ότι αυτό μπορεί να δώσει δώσει ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη και για την, ε, ε, να συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στο καταστατικό. Όσον αφορά την ψηφιακή επανάσταση και τις νέες ανάγκες, ε, τονίζεται ένας νέος τομέας στην τροπολογία 83 σχετικά με την ψηφιακή κοινωνία και ελπίζουμε να μπορείτε να υποστηρίξετε αυτή την τροπολογία που μιλάει για τον τομέα των μέσων ενημέρωσης όπου θα μπορούσαν οι εκδοτικοί εκεί να λειτουργήσουν ως συνεταιριστικές εταιρείε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά σας και η κυρία Χίρους λέει ότι ελπίζω ότι θα συνεχίσετε την καλή καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Κυρία Στάινουκ. Η κυρία Ρέγνερ μου ζήτησε να μιλήσω και για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και να διαβάσω την ε, παρέμβασή της ε, στο πλαίσιο των μελετών ε, που έχουν γίνει από την Επιτροπή για το Καταστατικό έχουν το στόχο οι τροπολογίες της ε, να εξετάσουν ε, αυτή την πρόταση της Επιτροπής που και πάλι δεν αφορά ε, αναδιατύπωση. Μιλάμε για σωστή εταιρική διακυβέρνηση και για σωστό συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο, για τα οποία πρέπει η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις ο λόγος για τον οποίο μέχρι τώρα υπάρχουν πολύ λίγες συνεταιριστικές εταιρείε δεν οφείλεται στην οδηγία, οφείλεται ε, στο ότι είναι πολύπλοκο το καταστατικό και ε, πολύ συχνά χρειάζεται να προσφεύγουμε στο εθνικό δίκαιο. Έχουμε 27 ε, διαφορετικά μοντέλα συνεταιριστικών επιχειρήσεων και σε ένα τέτοιο συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να δούμε πόσο πρέπει να ε, προωθήσουμε τις τροπολογίες που υπάρχουν στην ε, οδηγία. Ε, η κυρία Ρέγκνα θα συμμετάσχει στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών και επιπλέον χαίρεται για την πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. If there's no... Σα ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει άλλο σχόλιο, θα δώσω ξανά το λόγο στον εισηγητή Σβέν Γκίγκολντα. Συγγνώμη, διακόπτη η πρόεδρος. Δίνει το λόγο στον κύριο Μάν. Η πρόεδρος δεν κοιτάζει καθόλου αριστερά. Εσείς προς τα δεξιά, η πρόεδρος προς τα αριστερά δεν κοιτάζει. Αλλά πάντοτε χαίρομαι όταν προεδρεύετε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Σβέν ε, για τη συνεργασία που είχαμε σχετικά με το σημαντικό αυτό τομέα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το μοντέλο του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού. Είναι ένα, ένας καινούριο τομέας ε, και θέλουμε να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προτάσεις ε, και θέλουμε να επικεντρωθούμε στα πιο σημαντικά σημεία το 2012 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, αυτή τη χρονιά ε, για να επεξεργαστούμε αυτό το θέμα, γιατί τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ορίσει το 2012 ως Διεθνές Έτος ε, Συνεταιριστικών Εταιριών, Συνεταιρισμών. Θέλουμε να έχουμε καλές εμπειρίες από τα κράτη-μέλη, καλές ιδέες, να τα συνδυάσουμε όλα αυτά για να μπορούμε να κάνουμε κάτι προς όφελος και των μετόχων και των εργαζομένων όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε να λειτουργήσουν καλύτερα. Δεν έχουμε ακόμη μεγάλη εμπειρία επί του θέματο. Ε, αυτό οφείλεται στο ότι ήταν πολύπλοκα αυτά που είχαμε και είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι απλούστερο. Μπορούμε να έχουμε τι κατάλληλε διαρθρώσει ε, που θα μπορέσουν να εφαρμοστούν στην πράξη. Και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία ε, να δώσουμε σημασία και στις περιοχές της Υπέθρου, γιατί και εδώ έχουμε πολύ καλές εμπειρίες, τις οποίες μπορούμε ε, να μεταφέρουμε και σε άλλους. Από την εμπειρία μας αυτή μπορούμε να υποφεληθούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά σίγουρα και στην ε, συνάντηση των σκιωδών ε, εισηγητών μπορούμε να καταλήξουμε στις σωστές συμβαστικέ λύσεις, γιατί πρέπει να δώσουμε ένα σημαντικό μήνυμα προς τα έξω, ούτως ώστε να έχουμε τελικά αποτελέσματα τα οποία θα τιμούν την ε, κοινότητα. Σε πολλές χώρες δεν είναι καν γνωστή η έννοια των συνεταιριστικών εταιριών. Θα έχουμε λοιπόν μια κατάσταση από την οποία θα υποφεληθούν όλοι και πιστεύω ότι μόνο θετικά θα είναι τα αποτελέσματα. Σα εύχομαι καλή επιτυχία στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών και σα ευχαριστώ για την καλή μα συνεργασία. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο, ε, και ξαναδίνω το λόγο στον Σβέν Γκίγκολτ, αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Ευχαριστώ. Και μετά την παρέμβαση αυτή δεν νομίζω ότι γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό το θέμα, γιατί δεν είχαμε και μεγάλε διαφωνίε όσον αφορά ε, τι τροπολογίε. Με τι τροπολογίε τη Νάντια συμφωνώ, συμφωνώ με όλε και με τις δικές σας τροπολογίες, ε, λέει προς τον κύριο Μάνο, ο κύριος Κίγκολ. Ε, μερικές φορές υπήρχαν τροπολογίες για το ίδιο άρθρο. Όταν υπάρχουν πολλές τροπολογίες για το ίδιο σημείο, τότε πρέπει να βρούμε μια συμβαστική λύση, αλλά νομίζω ότι αύριο στη συνάντηση ε, των σχεδόν εισηγητών, των σχεδόν εισηγητών θα μπορέσουμε να τα ρυθμίσουμε. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ όλων των σχεδόν και βέβαια συμφωνώ και με τις παρατηρήσεις που κάνετε εκ μέρους της Εύελιν το κύριο πρόβλημα είναι το καταστατικό και δεν είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό μεταρρύθμιση. Πάντως το πολιτικό πλαίσιο αυτής της έκθεσης ε, βρίσκεται στην ενίσχυση ε, των συμπληρωματικών μέτρων για να ενισχύσουμε τις συνεταιριστικές εταιρείες και μάλιστα επειδή υπάρχει το 2012 ως Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών. Το μόνο πρόβλημα που είχα με τις τροπολογίες είναι ότι κάποιες τροπολογίες προσπαθούσαν ε, ε, να βάλουν την κοινωνική οικονομία κάτω από την ε, κοινή αγορά. Αυτή τη λογική δεν μπορώ να την ακολουθήσω. Η κοινωνική οικονομία είναι τμήμα της κοινής αγοράς, αλλά όχι υποδέστερο και σε ορισμένε τροπολογίε χρειάζεται να αλλάξουμε κάπως τη διατύπωση. Επίση, υπήρχαν κάποιε τροπολογίε ε, που ε, ε, λένε ότι λόγω της καπιταλιστικής μορφής της οικονομίας μας αυτές οι εταιρείε θα μοιάζουν πάρα πολύ με όλες τις άλλες επιχειρήσεις και αυτή είναι μια γενική ιδέα την οποία δεν ήθελα να τονίζουμε στην έκθεση. Αυτές είναι οι τροπολογίες που μου δημιουργούσαν κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν ήταν τροπολογίες που προτάθηκαν από τους ομιλήσαντες, άρα δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τώρα. Θα κάνουμε τη συνάντηση των σκιωδών και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Έχω προτείνει και εγώ κάποιες συμβαστικές τροπολογίες για να συμπεριλάβουμε ε, τις ιδέες όλων. Ελπίζω λοιπόν ότι θα υπάρχει συνένεση για την έκθεση αυτή και ευχαριστώ όλους για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Και για να αναφέρω και τις ημερομηνίε 22 ε, Νοεμβρίου ε, η συνάντηση της τροπολογίας, 23 ε, στην Επιτροπή Απασχόλησης Ψηφοφορία, 21 και 22 στις Επιτροπές Ζούρι και Γυναικών. Και πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο, θέλω να σας πω ότι συμφωνήσαμε με τους συντονιστέ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε την ψηφοφορία νωρίτερα, παραμένει η ψηφοφορία στις 5.30. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα κάνουμε ένα διάλειμμα όταν τελειώσουμε το επόμενο σημείο μέχρι να ψηφίσουμε στις 5 και 30. Όλε Κρίστανσεν είναι εισηγητής για το ενωσιακό πλαίσιο εταιρική διακυβέρνησης. Αλλά νομίζω ότι αντικαθίσταται. Mr. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όντω. μιλώ εξ ονόματος του συναδέλφου Όλε Κρίστενσεν. Μου δώσε ένα σημείωμα τώρα και μου λένε ότι έχει καθυστέρηση το αεροπλάνο του στο αεροδρόμιο της Κοπεχάγης. Από ό,τι φαίνεται στο επόμενο ημίωρο δεν πρόκειται να έρθει. Θα προσπαθήσω να σας τα πω εγώ σύντομα, γενικά ποια είναι η προσέγγιση των σοσιαλιστών και του Όλε Κρίστενσεν και η πρώτη μας αντίδραση επέναντι στις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Όπως γνωρίζετε, η έκθεση αυτή είναι σχετικά σημαντική. Πρόκειται από πλευράς Επιτροπής Απασχόλησης για την εισαγωγή κάποιων κριτηρίων που θα οδηγήσουν σε καλύτερη αποτελεσματικότητα γιατί είναι και χρήσιμο και απαραίτητο. Και πάντα θα πρέπει να υπάρχει μια εταιρική διακυβέρνηση όπου να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι. Να είναι οι εταιρείε μας έτσι ώστε το κεφάλαιο ε, να έχει ε, συμμετόχους τους ίδιους τους εργαζομένους. Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ε, επιχειρήσεων και το ευρωπαϊκό μοντέλο είναι το πιο αποτελεσματικό γιατί μέχρι σήμερα ακριβώς λειτουργεί γιατί συμμετέχουν στη διακυβέρνηση της εταιρεία οι εργαζόμενοι. Η δεύτερη κεντρική ιδέα του Όλε Κρίστασεν είναι ότι η διαφάνεια και ε, η ε, χρηστή διαχείριση είναι κάτι το οποίο είναι υπέρ των επιχειρήσεων. 71 τροπολογίες έχουν καταδεθεί και πρέπει να πω καταρχήν ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον της Επιτροπής μας. Γιατί η προοπτική απασχόλησης βεβαίως λαμβάνεται υπόψη και επίσης θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα και δεν θα είναι εύκολη η διαπραγμάτευση. Ωστόσο, οι περισσότερες τροπολογίες βρίσκουν είτε σύμφωνο τον Κρίστεσεν είτε πρόθυμο να διαπραγματευτεί. Γιατί είναι πολλέ τροπολογίε που αναφέρονται στι ίδιε παραγράφου με διαφορετική διατύπωση. Θεωρεί ο εισηγητή ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο συμφωνία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Γιατί στη συντριπτική του πλειονότητα οι 71 τροπολογίε είναι θετικέ και θέλουν να βελτιώσουν και να διευκρινίσουν την πρόταση. Ο εισηγητή λοιπόν θα έρθει σε επαφή τούτη τη βδομάδα με όλου του σκιώδει και θα προσπαθήσει να βρει όσο γίνεται περισσότερου συμβιβασμού, έτσι ώστε η έκθεση αυτή να είναι οριζόντια, εγκάρσια όπω τη λέμε και να έχει την καταπλειοψηφία υποστήριξη τη Επιτροπής μα. Όπω επίση είναι προφανέ, λέει στο σημείωμά του ο εισηγητή, ότι ορισμένε τροπολογίε που προσπαθούν να αποκλείσουν ριζικά ε, ορισμένα πράγματα, όχι να βελτιώσουν ε, τι σχέσει να είναι πιο γενικό το όραμα, πάντα προσπαθούν να καταστρέψουν αυτές τις ιδέες συμμετοχή των εργαζομένων και στη διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι ο εισηγητή δεν μπορεί να τι δεχτεί, ούτε να τι στηρίξει, ούτε να τι διαπραγματευτεί, γιατί θέλουν να μειώσουν τα δικαιώματα και να μειώσουν και την έκθεση και να την ξεδοντιάσουν. να μην έχει κανένα θένος, καμία δύναμη, κανένα κύρωση έκθεση. Λοιπόν, η πρώτη εντύπωση είναι ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ όλων, επικοδομητικό πνεύμα, συμβαστικές τροπολογίες. Θα σας τα πει και ο εισηγητής κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για να είναι όσο γίνεται ευρύτερη υποστήριξη και συνένεση στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι η ψηφοφορία είναι στις 5 παρατέταρτο. Έκανα λάθος εγώ γιατί ήταν ένα λάθος στα έγγραφά μου. 5 παρατέταρτο προβλέπεται να γίνει η ψηφοφορία και δεν αλλάζει. Άλλος κανείς? Ευχαριστώ, ο κύριος Ντεμπάκερ. Όπως μόλις ακούσατε, κάναμε και κάποιες τροπολογίες εμείς από την ομάδα μας εγώ προσβλέπω βεβαίω τη συνεργασία με τον εισηγητή και του διαφόρου και όλου εισηγητέ, έτσι ώστε οι τροπολογίε αυτέ να συζητηθούν σε επικοδομητικό πνεύμα. Εγώ κοίταξα όλε τι τροπολογίε, όπω υποθέτω κάνουν και ο εισηγητή και οι άλλοι σκιώδει. Θα χρειαστεί δουλειά ακόμα για να συγκεράσουμε και να συμφιλειώσουμε τι διάφορε θέσει, ε, γιατί θα χρειαστεί συμβιβασμό όντω για πολλά σημεία. Το πρώτο που θέλω να πω μας ενδιαφέρει είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια δεσμευτική νομοθεσία και κάποιες εθελοντικές συμφωνίες ή κώδικες συμπεριφοράς και δεντολογίας που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες. Σας παραπέμπω ιδιαίτερα σε ένα ε, γενικό θέμα μιας γενικής αρχής comply and explain ότι θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες και να εξηγούνται. Αλλά όλα αυτά είναι θέματα της επιχείρησης. Η ε, δεσμευτική νομοθεσία βεβαίως αφορά ε, κάποιες επιχειρήσεις, αν είναι μικρές, μικρομεσαίες και όχι εισηγμένες, είναι υπερβολικό να έχουμε δεσμευτική νομοθεσία. Μπορούν οι εταιρείε να συμφωνούν, να συνεννοούνται, αλλά όσο καλέ και προθέσει να έχουμε, δεν μπορούμε να καταπνίγουμε τι εταιρείε, να τι οδηγούμε σε κάποια ασφυξία. Καλή χρηστή διακυβέρνηση προωθείται σε όλες τις χώρες, αλλά το περιεχόμενο είναι ευέλικτο, ανάλογα ε, με την εταιρεία και τις μελλοντικέ της ανάγκες με βάση την ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που θα πρέπει να δούμε στο συμβιβασμό, το δεσμευτικό σε σχέση με την εθελοντική συμφωνία. Το δεύτερο, μια αηφόρο πολιτική ε, μισθών. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να καταργηθούν οι δυνατότητες ε, ε, αμοιβή των εργαζομένων με μετοχέ ή με, με, μερίδια ή με μερίσματα. Το θέμα του management τη διαχείριση εταιρεία δεν μπορούμε να το ορίζουμε εμεί. Είναι θέμα τη εταιρεία τη ίδια. Επίση, διαφάνεια. μπορεί να προσθεθεί ε, στη Γενική Συνέλευση ε, και μια έκθεση για την αμοιβή των εργαζομένων, για τη μισθολογία τους ή για τα ε, θέματα των μετοχών. Και κάποια άλλα θέματα που αξίζουν την προσοχή μας στην παρούσα έκθεση. Δεν μπορούμε να έχουμε one size fits all, δηλαδή μια λύση για όλους. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά των μικρών επιχειρήσεων, των οικογενειακών επιχειρήσεων που δεν είναι εισηγμένε στα χρηματιστήρια. Αυτά δεν μπορούμε να το βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην παρακολούθηση των διαφόρων καταστάσεων και συμβουλών και συστάσεων στα κράτη-μέλη. Και εγώ είμαι μεγάλος υπέρμαχος των ανταλλαγών, της ανταλλαγής μάλλον ε, βέλτιστων πρακτικών. Υπάρχει εμπειρία στα διάφορα κράτη ανάλογα με την εταιρεία ε, έχουμε μια προσέγγιση μιας ταχύτητας, δύο ταχυτήτων, ε, μια προσέγγιση που κοιτάει περισσότερο τη συμμετοχή των ενεχομένων, τη συμμετοχή ε, των μετόχων shareholders και shareholders stakeholders, συγγνώμη. Ε, πάντως αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην καταπνίξουμε τις εταιρείες, να μην τις εμποδίσουμε να λειτουργούν, πάντα με επικοδομητικό πνεύμα και συνεργασία και θα τα βρούμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέρκας, αν δεν έχει κανένας άλλος ε, να πει τίποτα. Μάλιστα. Αυτά που είπε ο κύριος Ντεμπάκερ δείχνουν με μεγάλη σαφήνεια ακριβώς τα σημεία που έχουμε συμφωνία και τις πιθανές τριβές που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στη συνεδρίαση των οδών εισηγητών με τον κύριο Κρίστενσεν. Χαίρομαι που όλα τα θέματα της διαφάνειας ή όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εταιρική διακυβέρνηση, τον κώδικα δεντολογίας και τον εθελοντικό μας βρίσκουν σύμφωνους. Οπότε πιστεύω ότι θα βρούμε σημεία σύγκλησης. Τώρα θα καταλάβει ο κύριος Ντεμπάκερ ότι εάν ο ίδιος είναι τελείως αντίθετος με οποιαδήποτε νομοθεσία, έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Κρίστενσεν θα σας παραπέμψει σε άλλες χώρες που υπάρχει νομοθεσία. Ο κύριος ε, ε, Ντεμπάκερ λέει ότι δεν είναι απλώς κρίσιμο αυτό το θέμα, αλλά ότι είμαστε πάρα πολύ επικριτικοί απέναντι. Θα πρέπει να ψάξουμε συμβιβασμούς κάπου στη μέση του δρόμου όχι να θέλει ο καθένας να επιβάλλει τη θέση του και να το παρατραβήξει. Δεν μπορούμε να μειώνουμε, να απαξιώνουμε οποιαδήποτε μορφή νομοθεσία, αλλιώ θα είναι πολύ δύσκολο να ε, βρούμε συνένεση. Να αναζητήσουμε ένα δρόμο με ευελιξία, με συνεργασία, με κανόνες και πάλι ευέλικτου ε, που να προσαρμόζονται ανάλογα με την κατάσταση. Γιατί πάρα πολύ συχνά εδώ στο Κοινοβούλιο, σε αυτή τη συζήτηση και σε άλλε. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη φιλοσοφία ότι η μεγαλύτερη ευελιξία είναι παντελής έλλειψη κανόνων. Όχι, έλλειψη κανόνων δεν είναι ευελιξία, είναι έλλειψη κανόνων. Ευελιξία είναι να έχει κανόνε, αλλά να εφαρμόζονται με τρόπο εύκαμπτο, όχι άκαμπτο, ανάλογα με την κατάσταση, με την εταιρεία κτλ. Οπότε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορούμε να συμφωνήσουμε και σε αυτά τα πιο επίμαχα, πάντα με πνεύμα συνεργασία και δεν θα πρέπει η ομάδα του κυρίου Ντεμπάκερ να θέλει να τραβήξει το σκηνή. Ευχαριστώ. Στην Επιτροπή 22 Νοεμβρίου θα το συζητήσουμε, στις 5 Δεκεμβρίου θα το εγκρίνουμε, στη Νομική Επιτροπή 20 Δεκεμβρίου που είναι αρμόδια από τις ουσίας και στην Ολομέλεια το Μάρτιο. Εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη, αλλά πρέπει να περιμένουμε για την ψηφοφορία. Διακόπτουμε τώρα μέχρι τις 5 παρατέταρτο για ε, να ψηφίσουμε. Παρακαλώ να φέρετε όλοι τις κάρτες σας, είναι δηλαδή 14 και 45 ακριβώς ψηφίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. σε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 Uh, uh, Καθίστε παρακαλώ, θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν έχετε λοιπόν τις κάρτες σας, βάλτε τις, βάλτε στις σχισμές για να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία της έκθεσης της Σιλβάνα Ράπτη. Πρώτη τροπολογία επί της οποίας ψηφίζουμε είναι η συμβιβαστική γάμα. Συμβιβαστική γάμα, ποια είναι υπέρ. Συμβιβαστική γάμα υπέρ. Um, those against. Κατά. That is carried. Εγκρίνεται. Προχωράμε λοιπόν. Uh, compromise, uh, we go down to amendment compatible with amendment 13. No. 18. Uh, Περνάμε στην τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Uh, 34. Those in favor. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Uh, 36. 37. 37 oral amendment. 37 με προφορική τροπολογία. Yeah. Ε, θα θέλαμε να προσθέσουμε στην τροπολογία 37, εκεί που αναφέρεται that the minimum weight, ότι το μήνυμο ημερομίσθιο προσθέτουμε according to national σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές. Are there objections to... Υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτή την προφορική τροπολογία. Ωραία, λοιπόν, ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 καταπίπτει συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 43 έχουν καταπέσει 44 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 45 uh, Close the vote. And 18... Τέλος ψηφοφορίας 18 υπέρ εγκρίνεται. 18 uh, υπέρ 10 κατά. Καμιά απόχη εγκρίνεται. 46. Είναι συμβατή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 καταπίπτει. 48 έχει αποσυρθεί. Και συμβαστική G υπέρ κατά. Αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά για τη συμβιβαστική G.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 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 58 είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 60 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε για την 60. Vote is closed. 20 in υπέρ, 14 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Α, όχι, συγγνώμη, πίπτη 63. Και 65 και 66. Χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα της 66 ψηφίζουμε. Υπέρ ποιοι είναι. Κατά. Αρχίζουμε τον έλεγχο για το πρώτο τμήμα της 66. Vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. 17-17 καταπίπτει. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. The vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. 31 in favor. 31 υπέρ, 3 κατά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κυρία εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία. Για το σχέδιο γνωμοδότης της κυρίας Ρέγνε. Διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικέ και εμπορικέ υποθέσει. Τροπολογία 10. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Άρθρο 19, σημείο 2, τροπολογία 11 της κυρίας Πάξας. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12, Τόμας Χέντελ, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Για την 12, τροπολογία 12. Le vote est ouvert. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 15 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Άρθρο 19, τροπολογία 3 της συγγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 13, Τόμας Χέντελ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 της εισηγήτριας Απεσύρθη. Τροπολογία 5 δεν είναι αποδεκτή. Τροπολογία 14 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το επαληθεύσουμε για την τροπολογία 14. Ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορία 20 υπέρ 15 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 15 της κυρίας Όμεν Ρόιτεν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Α, να επαληθεύσουμε τη 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. 15 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται όντω. Τροπολογία 7 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υπέρ, επαναλαμβάνουμε υπέρ τη 7. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε για την τροπολογία 8. Εψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 14 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 είναι μη παραδεκτή. Ξέχασα την 8. Τροπολογία 8 της εισηγήτριας υπέρ. Α, την ψηφίσαμε, δεν την ξέχασα. Την ψηφίσαμε. Λοιπόν, μετά την αιτιολογική σκέψη 1, τροπολογία 1 της εισηγήτριας. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 της κυρίας Παξά υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. 25 15 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώσαμε τις εργασίες μας. Ραντεβού στις 22 Νοεμβρίου για την επόμενη συνεδρίαση. Γνωρίζετε βεβαίως ότι στις 23 το απόγευμα Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση. Κυρία Λίν, ε, διαδικαστικό. Ναι. Αποφάσισα ότι τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου θα παραιτηθώ. Και το λέω, το ανακοινώνω ότι η τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου θα εγκαταλείψω το Κοινοβούλιο. Σας ενημερώνω στην Επιτροπή Απασχόλησης. Nous sommes très Κυρία Λίν, Μα συγκινεί ότι για πρώτη φορά το λέτε εδώ ενώπιό μας, είδα τα μέσα συναντήρωση των μελών της Επιτροπής για την αποχώρησή σας. Λυπούνται που δεν θα σας έχουν πια ως συνάδελφο και φαντάζομαι ότι για να λάβετε αυτή την απόφαση, ε, πλήρη γνώση και σοφία, θα έχουμε την ευκαιρία να σας αποχαιρετήσουμε σε άλλες περιστάσεις. Έτσι. Ε, φιλία και όπως αρμόζει μετά από την καλή συνεργασία που είχαμε εδώ στην Επιτροπή που υπηρετήσατε δεν απατώμε καθόλου τη διάρκεια της θητείας σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Έχουμε αυτή την ανακοίνωση. Λοιπόν, φεύγει η κυρία Λίνη τέλη Ιανουαρίου. Voilà une démonstration comme... Ιδού η απόδειξη ότι η φιλία και τα, οι ενδείξει αλληλεγγύη υπάρχουν. Μπορεί πολιτικά να είμαστε αντίπαλοι ε, και <laughs> μάλιστα στενάρα. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ. Τα ξαναλέμε στι 22 Νοεμβρίου. Συντονιστέ παραμένουν, παρακαλώ, στην αίθουσα αυτή. Στις 6.30 όμως.